Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τη συνεδρίαση της ομάδας μας. Επόμενο θέμα σε μέση διάταξη της Επιτροπής μας, η μελέτη κατόπιν ανάθεσης από το θεματικό τμήμα Β για να καταλάβουμε το θέμα καλύτερα του κανονιστικού υπερθεματισμού στα ευρωπαϊκά διαρθωτικά και επενδυτικά ταμεία. Τα πέντε διαρθωτικά και επενδυτικά ταμεία μετά από ε, την προκήρυξη διαγωνισμού, το θεματικό τμήμα Β που μας υποστηρίζει, ε, ζήτησε από την εταιρεία Spatial Foresight να εκπονήσει την παρούσα μελέτη η οποία μας παρέχει μια πλήρια και εξαντλητική ανάλυση των βασικών κανόνων, μάλλον των βασικών αιτίων ε, του κανονιστικού υπερθεματισμού και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να μειωθεί ή να ε, αποφεύγεται αυτός ο υπερθεματισμός των κανονισμών. Έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε τον κύριο Κάι Μπέμε, ερευνητή στο Spatial ε, Foresight, που θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που επιθυμούν να κάνουν ερωτήσεις ή σχόλια. Έχετε το λόγο αγαπητέ κύριε Μπέμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλό απόγευμα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση προσπαθήσω να σας δώσω μια γενική ε, εικόνα της ε, μελέτης μας ξεκινώντας από τον στόχο της μελέτης και τη μεθοδολογία της. Πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο ορισμός του κανονισμού, κανονιστικού υπερθεματισμού. Cold plating. Στο πλαίσιο του, των α, ταμείων και, του ε, και, και των επενδυτικών ταμείων, μετά θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά σε ποια σημεία του κύκλου προγραμματισμού εμφανίζεται αυτός ο κανονιστικός υπερθερματισμός και έπειτα θα δούμε ποιοι είναι οι λόγοι ποια είναι τα που οδηγούν σε αυτόν, ποια είναι τα αποτελέσματά του και θα οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα και συστάσεις. Ποιο ήταν ο στόχο λοιπόν αυτή τη μελέτη, Εξετάσαμε και τα πέντε διαφορετικά και επενδυτικά ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώντα να εντοπίσουμε περιπτώσεις κανονιστικού υπερθεματισμού, να δούμε τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και να σκεφτούμε τρόπους ε, αντιμετώπισης του προβλήματος, επίλυσης του προβλήματος. Προσπαθήσαμε με άλλα λόγια να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα πιο συστηματικά, γιατί ο κανονιστικός υπερθεματισμός δεν είναι το αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου κανόνα ή κανονισμού, αλλά ε, μιας γενικότερης προσέγγισης απέναντι στους κανόνες. Γι' αυτό χρειάζεται και μια πιο συστηματική προσέγγιση. Ε, ψηλέξαμε βιβλιογραφία και μελέτες, διοργανώσαμε συνεντεύξει με υπαλλήλους ευρωπαϊκών οργάνων, με τους δικαιούχους. Δημιουργήσαμε επίσης και ομάδες εργασίας, focus group, για να συζητήσουμε πιο αναλυτικά τα συμπεράσματα, προσπαθώντας να έχουμε ε, εκπροσώπηση και των 28 κρατών μελών, για να αντιληφθούμε πώς εκδηλώνεται το πρόβλημα στο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταφέραμε να καλύψουμε και τα 28 κράτη-μέλη. Ε, λιγότερο μάλλον περισσότερο καταφέραμε να ασχοληθούμε με 9, αλλά έτσι και αλλιώς ο στόχο της μελέτης δεν ήταν να συγκρίνουμε τα κράτη-μέλη μεταξύ του. Αναζητούσαμε παραδείγματα από κάθε κράτο μέλο. Πάντω, σα το λέω αυτό για να σα εξηγήσω ότι υπάρχει μια γενικότερη κάλυψη των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται να αναφερθώ μόνο σε ένα-δύο παραδείγματα. α πω συγκεκριμένα κράτη. Θα ήθελα να κρατήσουμε ε, στο μυαλό μας τέσσερις βασικούς όρους. Πρώτα απ' όλα ο ενεργός κανονιστικός υπερθερματισμός, active plating. Αυτό αναφέρεται στην δημιουργία διαδικασιών ή δημιουργία ε, υπρόσθετων υποχρεώσεων πέραν εκείνων που θεσπίζονται από τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ή επενδυτικών ταμείων. Δηλαδή, την ε, ενεργητική προσθήκη περισσότερων προϋποθέσεων. Όμως υπάρχει και ένας παθητικός, αν θέλετε, κανονιστικός υπερθεματισμός, δηλαδή όταν υπάρχει η δυνατότητα ε, τα πράγματα να γίνονται πιο απλά και δεν την αξιοποιούμε. Ενώ θα μπορούσαν δηλαδή να γίνονται με λιγότερη γραφειοκρατία, με λιγότερο κόστος, ε, δεν αξιοποιούμε αυτή την ευκαιρία, δεν την εκμεταλλευόμαστε. Μετά, ένας επιπλέον όρος που μας ενδιαφέρει είναι τα, το διοικητικό κόστος. Είναι εκείνο που επομίζεται το κράτος μέλος που υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα και την πολιτική συνοχή και το διαχειριστικό άχθος είναι το κόστος και οι διαδικασίες επιπλέον που αναγκάζεται ο δικαιούχος να δημιουργήσει και να επομιστεί. Σας ζητώ να ε, ε, θυμάστε αυτούς τους τέσσερις όρους γιατί θα αναφέρομαι σε αυτούς κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου. Στο διάγραμμα που βλέπετε στην οθόνη σας και το οποίο μπορείτε να δείτε και στην έκθεση, στα αριστερά έχουμε το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πρέπει και να ακολουθήσει κανείς εάν θέλει να διαχειριστεί κονδύλια από διαρθρωτικά ή επενδυτικά ταμεία. Και μετά, με τα κίτρινα βελάκια, ε, εμφανίζονται οι επιπλέον ε, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που πηγάζουν από άλλα, άλλους κανονισμούς, άλλα πλαίσια, εθνικά ή ευρωπαϊκά. Και επιπροσθέτως, το κίτρινο μεγάλο βελάκι στα δεξιά είναι για το ζήτημα της ερμηνείας. Αυτό που αποφασίζει να κάνει μια δημόσια αρχή όταν απαντάει δεν ξέρω τι να σας πω τώρα, τι να κάνουμε με αυτό και, και επιλέγει την πιο περίπλοκη λύση. δημιουργώντας επιπλέον κόστος στο επίπεδο της διαχείρισης και της υλοποίησης του προγράμματος και περι, περαιτέρω γραφειοκρατία το οποίο βέβαια έχει ω αποτέλεσμα αύξηση του κόστους και για τον τελικό δικαιούχο, γιατί του ζητάμε να κάνει παραπάνω πράγματα. Προσπαθούμε με αυτό το διάγραμμα να δείξουμε ότι οι διάφορες αυτές επιλογές έχουν προσθετικό ε, χαρακτήρα. σε οποιοδήποτε στάδιο της υλοποίησης του προγράμματος, σε οποιοδήποτε σημείο του κύκλου προγραμματισμού, μπορεί κανείς να εντοπίσει περιπτώσεις κανονιστικού υπερθεματισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν εθνικοί κανόνες ε, που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ανατίθενται ε, ερμοδιότητες σε ενδιάμεσες αρχές δημιουργούν τέτοιον υπερθεματισμό. Ή μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο επίπεδο της διαχείρισης ενός συγκεκριμένου έργου, για παράδειγμα επιπλέον κριτήρια για την επιλεξιμότητα πέραν εκείνων που θεσπίζονται στο, στην νομοθεσία την Ευρωπαϊκή ή επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία ζητούνται και τα οποία πρέπει να ελέγχονται. Πολλές φορές ε, είναι δικαιολογητικά τα οποία είναι δύσκολο να αποκτήσει κανεί, είναι περίπλοκο να αποκτήσει κανεί και τα οποία δεν συνδέονται και άμεσα με την αίτηση χρηματοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να οδηγηθούμε σε υπερβολέ. Και στην έκθεσή μα, στην έκθεση που παρουσιάζει την μελέτη, θα δείτε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν έχω βέβαια χρόνο τώρα να μιλήσω για αυτά, αλλά αν σα ενδιαφέρει θα τα βρείτε στο, στο κείμενο. Περνάμε τώρα στο ζήτημα της παρακολούθηση και των υποβολή εκθέσεων. Ε, είναι κάποια στοιχεία, κάποια προβλήματα τα οποία έρχονται και ξανάρχονται από, και τα ακούμε από πολλά εμ, κράτη-μέλη και στο πλαίσιο πολλών διαφορετικών προγραμμάτων. Ε, το κυριότερο είναι η συχνότητα της υποβολής εκθέσεων. Ότι μας, μας λένε ότι μας ζητούν να υποβάλουμε εκθέσεις πολύ συχνά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη συνοχής ε, το, και η ασάφεια σε σχέση με το, τις εκθέσεις που ζητείτε να υποβάλλονται, μερικές φορές για θέματα τελείως άσχετα. Ή αν σκεφτεί κανείς πόσο πολύ χαρτούρα ζητείτε από τους δικαιούχους να υποβάλλουν για να ε, εκταμιευθεί ένα ποσό για να καλυφθεί μια δαπάνη σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι αυτό που ζητείται από τις δημόσιες αρχές ξεπερνάει κατά πολύ τις υποχρεώσεις που θα είχαν αυτές οι αρχές με βάση το νομικό πλαίσιο. Επίσης φαντάζομαι ότι πολλοί θα έχετε ακούσει και θα γνωρίζετε ότι εξαιτία των λογιστικών ελέγχων οδηγούμαστε σε υπερβολές, οδηγούμαστε σε προσεγγίσεις πολύ πιο ε, αυστηρές από ό,τι στην πραγματικότητα προβλέπονται στην νομοθεσία. Με επιπλέον κριτήρια, με επιπλέον προϋποθέσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώσαμε ο ε, οικονομικός έλεγχος, ο λογιστικός έλεγχος να ξεπερνάει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έπρεπε να κινείται. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και για τους διαχειριστές των προγραμμάτων, αλλά και για τους δικαιούχους. Και για τους ελεγκτές. Το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Ποιοι είναι οι λόγοι για τον κανονιστικό υπερθερματισμό. Γιατί φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ε, τι σημαίνει κανονιστικός υπερμαθηματισμός και από πού προέρχεται. Περισσότεροι νομίζουμε ότι είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας να καλύψουμε και άλλους στόχους πολιτικής. Αυτός είναι ένας, ένας από τους λόγους όμως. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί. Θα βρείτε παραδείγματα και στην έκθεση. Για παράδειγμα, οι αλλαγέ στους κανονισμούς, οι, οι στην υιοθέτηση νέων κανονισμών, που συχνά οδηγούν σε ασάφειες και εκεί ακριβώς αρχίζει ο κανονιστικός επερθεματισμός. Όταν υπάρχει ένα κενό και οι διάφορες δημόσιες αρχές αποφασίσουν να το καλύψουν η καθεμιά όπως νομίζει. Και αρχίζουν για να είναι καλυμμένοι να ζητούν ε, περισσότερα. Προτιμούν να ζητάνε περισσότερα από το να απλοποιήσουν τη διαδικασία. Ένα άλλος λόγος που οδηγεί σε κανονιστικό υπερθεσματισμό είναι παλαιότερες ε, άσχημε εμπειρίε. Δηλαδή ακούσαμε εκπροσώπους διαχειριστικών αρχών να μα λένε «Ε, είχαμε παλιά έναν λογιστικό έλεγχο, μας βρήκε προβλήματα και γι' αυτό από τότε ζητάμε. Αλλά ο... και επίσης δεν θα πρέπει να υποτιμούμε γεγονό ότι στι διάφορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διαφορετικέ νοοτροπίε όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση. Στι περισσότερε συνεντεύξεις πάντως αυτό που ακούσαμε ε, είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν εξαιτία του φόβου των ελεγκτών. Και συνολικά η πολυπλοκότητα του συστήματος είναι υψηλή. Ε, φάνηκε αυτό από τις ε, συνεντεύξεις και από το focus group και ταυτόχρονα φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένοι ε, παίκτες στο σύστημα, ορισμένοι από αυτούς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, που έχουν συμφέρον να καθιστούν το σύστημα περίπλοκο ε, ως έναν τρόπο για να διατηρούν την εξουσία τους ή για να φροντίζουν να καθυστερούν τα πράγματα. Προσθέτονται σε ένα επιπλέον βήμα, μια ακόμα υπογραφή κτλ. Και έτσι δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο, γιατί το σύστημα ήταν περίπλοκο από μόνο του. Υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να το κάνουν πιο περίπλοκο και ούτω καθεξή. Ποιε είναι οι επιπτώσει τώρα του κανονιστικού υπερθεματισμού στο επίπεδο του εθνικού και το διαχείριση των προγραμμάτων. Βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση του κόστου. όλο και περισσότεροι πόροι που θα ήταν διαθέσιμοι για τεχνική βοήθεια σπαταλώνται για αυτές τις διαδικασίες και δεν περισσεύουν μετά. Και τελικά ε, σπαταλούμε χρήματα χωρίς να υλοποιούμε τους, τα, τα, τα δαπανούμε για τους λόγους για τους οποίους τελικά έχουμε αυτές τις πολιτικές. Υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εξεταστεί μια αίτηση, για να δοθεί η απάντηση στον ετούντα. Και γενικά αργούν τα πράγματα. Και βεβαίως όσο πιο υψηλά ανεβαίνει κανείς στι διάφορε κλίμακε τη δημόσια διοίκηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιφυλακτικότητα, τόσο πιο πολύ φοβούνται οι υπάλληλοι να κάνουν λάθος για τι επιπτώσει που θα έχει. από τις διάφορες διοικητικές διαδικασίες, αυτό που φάνηκε από τις συζητήσεις που είχαμε, ήταν ότι κυρίως οι μικρότερη δικαιούχοι, μικρές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μικρές ε, δημόσιες αρχές, περιφέρειες ας πούμε, η δήμοι. Είναι αυτοί οι μικροί παίκτε οι οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή του του απαιτούμενου πόρου για να ανταποκριθούν σε όλη αυτή τη γραφειοκρατία και τελικά φοβούνται και δεν υποβάλλουν καν αίτηση. Άρα το, οι δυσμενείς επιπτώσεις του κανονιστικού υπερθεματισμού κλείτουν κυρίως τους μικρότερους. Εκείνοι είναι που πρώτοι θα σκεφτούν ε, να, να βρουν έναν άλλον τρόπο αντί να υποβάλουν αίτηση σε ένα τόσο περίπλοκο και γραφειοκρατικό πρόγραμμα που να βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά ήταν δύο τελευταίες διαφάνειες ε, για να έχουμε την πλήρη εικόνα και πώς ε, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ποιο είναι το σύστημα και ο τρόπος με τον οποίο ε, εισχωρεί το κανονιστικός υπερθεματισμός. Συμπεράσματα από δύο λόγια και αν ενδιαφέρεστε να βαθύνουμε στη συζήτηση. Γενικά ο κανονιστικός υπερθεματισμός αυξάνει το διοικητικό κόστος και άχθος. Αυτό το έχουμε δει. Και σύμφωνα με τις μελέτες είναι και υψηλό το ποσοστό. Και εδώ παίζουν ρόλο και οι δύο μορφές ενεργού και παθητικού, ενεργητικού μάλλον και παθητικού υπερθυματισμού. Και σε οποιαδήποτε διαδικασία τη διαχείριση. δεν είναι μόνο στο επίπεδο σχεδιασμού προγράμματος ή στο εθνικό επίπεδο ή στο τοπικό επίπεδο. Είναι σε όλο ε, τον κύκλο και όλη τη διάρκεια ζωή του ε, έργου. Επίσης, Μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ διαφόρων ταμείων και διαφόρων δραστηριοτήτων, υπάρχουν, αλλά δεν έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην ανάλυση μας. Ε, η διαφορά είναι περισσότερο μεταξύ κρατών μελών λόγω των διαφορετικών διοικητικών ε, νοοτροπιών που επικρατούν και ε, αντιλήψεων. Και συχνά το κίνητρο και ο λόγος ε, για τον υπερθεματισμό είναι ε, ε, φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Γιατί ε, ότι έχω υποστεί έλεγχο, λογιστικό, έχω βρει τον πελά μου και δεν θέλω να το ξαναβρω μπροστά μου. Γι' αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Ε, ταυτόχρονα είχαμε και συζητήσεις εάν ε, και κατά πόσο υπάρχουν περιπτώσεις που να είναι απαραίτητος ο υπερθυματισμός. Σε ορισμένε περιπτώσεις μπορεί να θεωρείται υπερβολή και σε άλλες ε, δικαιολογημένος, γιατί υπάρχει κάποιος λόγος. Ε, όταν βάζουμε επιπλέον στόχους ή συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εδώ θα πρέπει να σταθμίζονται διάφοροι στόχοι και ε, σκοποί. Παράδειγμα, ε, η πράσινη δημοπράτεση ε, ας πούμε, όταν προκυρήσω ένα έργο και θέλω και προστασία του περιβάλλοντος με συγκεκριμένο πράσινο τρόπο εντό εισαγωγικών, αυτό είναι μια επιπλέον κανονιστική ρύθμιση, αλλά ε, είναι προς όφελος του περιβάλλοντος ή είναι δικαιολογημένη γιατί επιδιώκουμε κάτι διαφορετικό. Και όπως σας είπα προηγουμένως, αυτό μπαίνει και στη συνδιαχείριση. μπορεί να σημαίνει ότι όλοι συμμετέχουν στα διάφορα επίπεδα. Επόμενες ε, διαφάνειες αφορούν τις ε, συστάσεις. Τι μας λένε λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι. Αν θέλετε να μειώσετε το ε, γραφειοκρατικό άχθος, ορίστε τι πρέπει να γίνει. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαφάνεια, ευκρίνεια, απλοποίηση και μην αλλάζετε συνέχεια τους κανόνες. Δεν πρόκειται ποτέ να είναι τέλειοι οι κανόνες, αλλά κάθε νέα αλλαγή δημιουργεί μια περίοδο αβεβαιότητας. Δηλαδή, ο κόσμος ζητάει σταθερότητα, συνέχεια, ε, ακόμα και αν θυσιαστούν ορισμένες μικρές βελτιώσεις. Σε εθνικό επίπεδο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ε, και η συνοχή Φτάνει. Και μην μας ζητάτε περισσότερο χαρτοβασίλειο. Και επίσης λάβετε υπόψη σα την οτροπία της δίκης κάθε χώρα, της κρατική μηχανή που δεν είναι όλες ίδιες. Σε επίπεδο προγράμματος θα πρέπει να δίνετε σαφήνεια στους δικαιούχου και ε, να γνωρίζουν περισσότερο και να κάνουν περισσότερη χρήση ε, ε, των διαδικασιών μειωμένου κόστου σε διάφορα επίπεδα χρειάζεται διάλογος και διάλογος με τους οικονομικούς ελεγκτές πολύ νωρίς έτσι ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι τι τους περιμένει, τι θέλουν οι ελεγκτές, τι θέλουν οι επιθεωρητές και δεν χρειάζεται κανείς να φοβάται ε, τον ευνίδιο έλεγχο ότι ξαφνικά μπορεί να εμφανιστεί ο επιθεωρητής και, και να τους φοβούνται χωρίς να τους έχουν συναντήσει και να έχουν συζητήσει μαζί τους. Απλώς φοβούνται την ιδέα ότι μπορεί να έρθει ο έλεγχος. Και θα πρέπει να δούμε αν τηρούμε τους κανόνες που ε, καταλήγουμε, ποια είναι η συμμόρφωση, ποια είναι η απόδοση και να ε, ε, χρησιμοποιούνται διαδικασίες μικρότερου κόστους. Τελευταία διαφάνεια, μας είπαν να κοιτάξουμε όχι μόνο το τρέχον σύστημα, αλλά τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Την πολιτική συνοχής δηλαδή μετά το 2020 να εξετάσουμε ποιες είναι οι βασικές ιδέες εκεί. Στη συζήτησή μας φάνηκε ξεκάθαρα από τους διάφορους ενεχομένους ότι θέλουν τρία διαφορετικά μοντέλα ε, για να μειωθεί ο κανονιστικός υπερθεματισμός. Το πρώτο ήταν να διατηρηθεί μεν το παρόν σύστημα, γιατί έχει μια σταθερότητα και έχει σημασία να μην αλλάζουμε συνέχεια και να προσπαθήσουμε λίγο να ξεφύγουμε από τη συμμόρφωση προς τις επιδόσεις ε, αυτό ε, μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί ε, το gold plating. Υπάρχουν και άλλοι που μας είπαν ότι θέλουν περισσότερους κανόνες και πιο αυστηρούς αν θέλουμε να μην φεύγουν τα κράτη-μέλη σε αυτό το εργαλείο του κανονιστικού υπερθεματισμού. Άρα να υπάρχει input, έλεγχος και μόρφωση. Και υπάρχουν και εκείνοι που μας είπαν ότι χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία και εμπιστοσύνη. Και πολλά κρατημέλη και πολλοί δικαιούχοι. Γιατί μας είπαν όσο περισσότερο μας ελέγχεται, τόσο αναποτελεσματικό είναι το σύστημα, ανενεργό και άκαμπτο. Και επικρατεί και μια δυσπιστία, μια καχυποψία. Δηλαδή υπάρχει ευελιξία και εμπιστοσύνη και το πρόγραμμα θα βγει με το σωστό τρόπο. Δεν χρειάζεται πια τους δρακόντιο έλεγχο, λέει η τρίτη εκδοχή. Θα πρέπει να εστιάζουμε στα επιτεύγματα, στις επιδόσεις, και όλα να έχουν γίνει φυσικά σύνομα, αλλά να μην είστε βολικά σχολαστικοί και ε, με νομικίστικο πνεύμα να ασχολείστε με τις λεπτομέρειες. Αυτά είναι τα τρία που μας πρότειναν οι ε, συμμετέχονται στο πρόγραμμα στη μελέτη. Εμείς δεν επιλέγουμε, απλώς σας αναφέρουμε ποια είναι ε, τα υπέρ, τα κατά ε, για τα διάφορα συστήματα, έτσι ώστε να ε, δώσουμε τροφή για συζήτηση. Δεν θέλω να πάρω πάρα πολύ από το χρόνο σας, θα σταματήσω εδώ και περιμένω και τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπόμ για αυτές τις πολύ διαφωτιστικές πληροφορίες. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πάρει το λόγο, να θέσει ερωτήσεις. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την ε, ε, μελέτη αυτή, πολύ σημαντική για μας. Είναι um, uh, μια καλή μέθοδος αυτή για να δούμε πώς απορροφώνται οι πόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την παρουσίαση αυτή διαπίστωσα ότι βρισκόμαστε ενώπιον μια αβεβαιότητας ερμηνείας των κανονισμών και ως εκ τούτου έχουμε ένα εφέ ντόμινο, φτάνουμε δηλαδή σε μια υπερβολη, σε υπερβολικό ρυθμιστικό πλαίσιο επειδή φοβόμαστε μήπως κάνουμε λάθος. Όμως εγώ ρωτώ γιατί δεν είναι δυνατόν ή μάλλον σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να ε, έχουμε μια μόνη ε, διαδικασία. Εσείς μιλήσατε για διαφορετικές νοοτροπίε από την διοικητική άποψη. Ναι, όντω. μπορούμε να το δεχτούμε αυτό ότι έχουμε διαφορετικές διοικητικέ ε, ε, νοοτροπίε και κουλτούρες, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην δέχεται μία απλοποιημένη ε, ενιαία διαδικασία που να είναι απόλυτα σύμμορφη προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να γνωρίζουμε δηλαδή ποιος είναι ο δικός χάρτης για τα κονδύλια και να γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει σε κάθε φάση. Και από αυτό πρέπει να επιμείνουμε, να υπάρχει μια ενιαία διαδικασία για όλα τα κράτη της Ένωσης. Εάν το καταφέρουμε αυτό θα μειώσουμε το διοικητικό κόστος, γιατί ακριβώς εσείς είπατε ότι εφόσον γίνονται πολλοί και διάφοροι έλεγχοι υπάρχει μια μεγαλύτερη ε, επιφυλακτικότητα όσον αφορά την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η υπερβολική λοιπόν νομοθεσία δημιουργεί φόβο, προκαλεί φόβο και σε αυτό το θέμα πρέπει να εργαστούμε. Μάλιστα, θα ακούσουμε πρώτα τις ερωτήσεις ε, και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις. Κόλτσακ, συνάδελφος Κόλτσακ. Η συζήτηση αυτή με ενδιαφέρει. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η εισήγησή σας. Η συνεργασία ανάμεσα σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή με επαγγελματικές οργανώσεις στον ε, δικαστικό τομέα όπου θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία, με κάνει να αναρωτηθώ κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να αποφύγουμε ακριβώς αυτό την συγκέντρωση περαιτέρω ρυθμίσεων και κανονισμών που θα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε μελετήσει λίγο το θέμα σε επίπεδο τσεχικής δημοκρατίας και διαπιστώσαμε ότι την τελευταία περίοδο, από το 2012 δηλαδή, Υπολογίζαμε πως το 1 τέταρτο των νέων υποχρεώσεων της ε, τσεχικής δημοκρατίας που αρχικά αιτιολογείται ακριβώς από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην ουσία συνδεόταν με τον ε, κανονιστικό υπερθεματισμό και μπορούμε ίσως εδώ να μιλήσουμε και για υποχρεώσεις ή καταστάσεις συγκεκριμένες στην Τσεχική Δημοκρατία όπου πραγματικά υπήρξε κάποιο αίτιο που συνδεόταν με το υπερθεματισμό και όχι αναγκαστικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας ε, στην Τσεχική Δημοκρατία. Ας πούμε, για παράδειγμα, με, όσον αφορά τις ε, μπαταρίες, δεν είναι πρόκειτο για ε, νέο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά για υπερθεματισμό. Ποια λύση λοιπόν διαβλέπετε για αυτό το πρόβλημα και έπειτα διερωτώμαθα κατά πόσο η εκτίμηση του αντικτύπου, δηλαδή μια ανάλυση όταν κάποιο κράτος μέλος υιοθετεί διατάξεις, πώς και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε λύση αυτού του προβλήματος. Γιατί πρέπει πάντοτε να μπορούμε να αποδείξουμε γιατί ένα συγκεκριμένο εθνικό όργανο θέλει να συμπεριλάβει συγκεκριμένες διατάξεις. Ε, κύριος Νίλσον, ευχαριστώ ε, για την παρουσίαση αυτής της μελέτης, η οποία μας περιγράφει κάτι που όλοι γνωρίζουμε ουσιαστικά πάρα πολύ καλά. Και καλό είναι που ε, μας παρουσιάσατε τη μελέτη αυτή, γιατί έχουμε έτσι τη συνολική εικόνα. Αναφερθήκατε λίγο και στον ε, ρόλο των ε, επιθεωρητών, των ε, οικονομικών ελεγκτών που προκαλούν κάποιο φόβο. Πέρα όμως από τους ελεγκτές υπάρχουν οι σχέσεις των εθνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εθνικές αρχές φοβούνται μήπως κάνουν κανένα λάθος και μήπως πάει κάτι στραβά και μήπως τους επιπλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό υπερβάλλουν καμιά φορά. Εν πάση περιπτώσει, η μελέτη αυτή θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τις μελλοντικές μας συζητήσεις σχετικά και έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστεί να επικεντρωθούμε περισσότερο στα αποτελέσματα, στις επιδόσεις. Πρέπει να βρούμε ένα σύστημα Έχω πολλά παραδείγματα, αν θέλετε να σας δώσω, όπου προσπάθησαν κάποιοι, αν μη τι άλλο, να απλουστεύσουν τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, σε κάποιες τουριστικές περιοχές προσπάθησαν να ομαδοποιήσουν κάποιες επιχειρήσεις, 100 επιχειρήσεις ας πούμε, ε, τουριστικές, με μια πλατφόρμα ε, έτσι ώστε να ε, διαχειρίζονται μεγάλα προγράμματα τουριστικού ενδιαφέροντος. Και χάρη λοιπόν σε αυτές τις πλατφόρμες μπορούν πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πρόγραμμα ή σε ένα μεγάλο έργο. Είναι λοιπόν στη διάθεση των μικρών επιχειρήσεων και ξέρουμε ε, ε, ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Θα μπορούσε να είναι αυτό ένα παράδειγμα για τα μεγάλα έργα υπέρ των μικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, όπου έχουμε πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, να δημιουργούνται τέτοιες πλατφόρμες επιδόσεων και αποδόσεων και να έχουν η ενδιαφερόμενη πρόσβαση. Λύσεις λοιπόν υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης και να μην επιμένουμε ε, στις διαδικασίες αλλά στα αποτελέσματα. Κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ αγαπητέ φίλε. Επιτρέψτε μου να μιλήσω ρουμανικά, διότι φαίνεται ε, ότι το έχουμε ξαναδεί αυτό. Είναι ε, μια έμονη ιδέα. Όλοι ε, λέμε θέλουμε απλούστευση και ακούμε ας έχουμε απλούστευση, ας προχωρήσουμε προς πιο εύκολη πρόσβαση στα κοινοτικά κονδύλια. Όσο τα λέμε αυτά, όσο περισσότερο, τόσο πιο περίπλοκη είναι η πραγματικότητα. It's a kind of Kafka. Αυτά είναι καταστάσεις τύπου Kafka και στρέφονται απέναντι και τουλάχιστον ε, σε αυτά που λέμε δημόσια ή στη δημόσια βούληση. Τώρα θα βάλω τα ρουμανικά γυαλιά για να μιλήσω στη γλώσσα μου και να σας αναφέρω τη ρουμανική πραγματικότητα. Ένα πρώτο λοιπόν ε, στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι το εξής. Και το λέει σωστά ε, το επισημένη η μελέτη. υπάρχει ένας πανικός που παραλύει όλα αυτά τα κριτήρια οικονομικού ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, τρομοκρατούν ε, τα κράτη-μέλη, ε, τα οποία φοβούνται τους ορκωτούς ε, ελεγκτές, τα ελεγκτικά συνέδρια. Ε, δεν ακολουθούν τους βασικούς κανόνες, δεν ακολουθούν τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, αλλά περιπλέκονται όλο και περισσότερο οι έλεγχοι. Και συχνά στις διάφορες γενικές διευθύνσεις δεν ακολουθούνται οι ίδιοι έλεγχοι με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Δεν είναι τυποποιημένες οι διαδικασίες ελέγχου. Στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που δεν ανταποκρίνονται απολύτως σε αυτά που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν θα ήταν πιο απλό να έχουμε νέους λογιστικούς ελέγχους, να έχουμε ευρωπαϊκούς και να ισχύουν παντού, εναρμονισμένα στα διάφορα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, είμαστε εντάξει. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Ρουμανία. Στο ελεγκτικό μας συνέδριο υπάρχουν κριτήρια που είναι πολύ πιο αυστηρά και πολύ πιο ε, ρακόντια. Και είναι και κατάχρηση, αν με ρωτήσετε. Ε, και δυσκολεύουν απίστευτα τη ζωή των δικαιούχων εκείνων που ζητούν ε, χρηματοδότηση. Ένα άλλο στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα πράγματα αυτά οι δικαστικές αρχές ε, με υποτιθέμενες ή ύποπτες περιπτώσεις απάτης. δεν υπάρχει μια εισαγγελία που να ακολουθεί τα ίδια κριτήρια. Α πούμε, όταν έχεις μια υποψία απάτης, θα θεωρούσε κανείς ότι είναι συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται παντού, ανεξαρτήτως ε, κράτους μέλους. Ε, λοιπόν, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στη Ρουμανία ε, η κατάσταση είναι πραγματικά τρομακτική. Έχουμε ένα σώμα καταπολέμησης της διαφθοράς που λέγεται DNA στη ε, ε, Ρουμανία. Ε, εγώ την υποστηρίζω. Προφανώς θα πρέπει να γίνεται σωστή και χρηστή διαχείριση των κονδυλίων, αλλά χρειαζόμαστε κοινή ερμηνεία και κοινή πρακτική στον τρόπο με τον οποίο επιβάλλουμε τον Ευρωπαϊκό Νόμο στην Ευρώπη. Και όχι ερμηνείες κατά το δοκούν ομαδικές και προσωπικές ανάλογα με τη χώρα. Φυσικά φοβούνται μετά ε, οι ε, πολίτες να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης. Αυτό οδηγεί σε πραγματική παράλυση. Είναι πραγματικότητα στη Ρουμανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα γνωρίζει όλα αυτά πάρα πολύ καλά. Και θα τολμούσα να πω ότι το ενθαρρύνουν κιόλα. Ένα τελευταίο που είπατε εσείς. Θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και να λέμε μέσα σε αυτό το διάστημα δεν πρόκειται να αλλάξει νομοθεσία για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ή να βάλουμε μια προθεσμία από τη στιγμή της έγκρισης του ΕΣΠΟ, ας πούμε, ε, δίνεται ένα διάστημα για να οριστούν οι κανόνες. Αλλά από εκεί και πέρα, μετά την εκνοή της προθεσμίας, δεν επιτρέπονται αλλαγές ε, στο νομικό πλαίσιο και στο θεσμικό πλαίσιο για να κανονίζει ο καθένας την πορεία του. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πέρυσι είχαμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα και στη συνέχεια έγιναν αλλαγές τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο για τους κανόνες που ισχύουν. Ε, τρελαίνεται μετά ο δικαιούχο. Δεν ξέρει ε, τι ισχύει, έχει ετοιμάσει την αίτησή του με βάση κάποιους κανόνες και όταν θέλει να το υποβάλει, του λένε «Α, ξέρεις, άλλαξε ο τάδε κανόνας». Το κάνει δεύτερη φορά, πληρώνει και κάτι παραπάνω, διοικητικό ε, κόστος και μετά του λέει «Α, ξέρεις, άλλαξε ξανά». Ε, δεν είναι αυτά πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα γνωρίζει, επαναλαμβάνω. Χρειαζόμαστε κάτι που να σταματήσει αυτή τη δημιουργικότητα, εν Γιατί και ε, αστάθεια ε, δημιουργεί αυτό και ε, αβεβαιότητα. Κάτι άλλο που τονίζει η μελέτη και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το διοικητικό κόστος αλλά και το οικονομικό κόστος που πλέον έχει καταντήσει αφόρητο ιδιαίτερα στους μικρομεσαίους ή και στις μικρομεσαίες ε, τοπικές αρχές, δήμους και κοινότητες. Σε πρώην βιομηχανικές περιοχές που είχαν ε, ε, μία και μοναδική παραγωγή σε πρώην κομμουνιστικά κράτη που είναι φτωχές περιφέρειες και δεν μπορούν να τρέχουν τόσο περίπλοκα προγράμματα δεν έχουν τους πόρους, δεν έχουν καν το λεξιλόγιο να καταλάβουν τι είναι τα ολοκληρωμένα προγράμματα που ε, ε, υποστηρίζονται από διάφορα ταμεία. Μετά, οι μικρομεσαίοι δεν θα πρέπει να συμμετέχουν. Αλλά όταν είναι να μπλέξουν τόσο άσχημα, σου λέει άστο καλύτερα, γιατί δεν θεωρούν ότι είναι σε θέση να το διεκπαιρεώσουν, ότι τους ξεπερνάει δεν θέλουμε να συμμετέχουν οι άνθρωποι αυτοί ε, στα διαρθρωτικά ταμεία. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει τη μελέτη αυτή και ε, θα σταματήσει αυτές τις πρακτικές. Σας είπα, είναι κάφκα αυτά ε, που έχουμε στα διαρθρωτικά ταμεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον να σε ακούμε πάντα, Βίκτορ. Ο συνάδελφος Βόν. Uh, Thanks, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Βίκτορ. Χρησιμοποιήστε τη λέξη συμπερασματικά. Κλείνω πέντε φορές. Όπως ε, είπε ο εκπρόσωπος της ε, εταιρείας μελετών, μας είπε ότι ήταν μια ανάλυση ε, υφιστάμενων μελετών, μια βιβλιογραφική μελέτη αυτή η έκθεση θα ήταν χρήσιμο να είχαμε ορισμένα πιο συγκεκριμένα παραδείγματα στη συζήτησή μας. Γιατί ε, πολλοί από εμάς γνωρίζουμε, βέβαια, έχουμε στο μυαλό μας συγκεκριμένα παραδείγματα όπως εκείνα που ε, αναφέρατε από τις περιφέρειές μας. Δόθησαν κάποιοι λόγοι που οδηγούν σε αυτόν τον κανονιστικό ε, παρθυματισμό, οι αλλαγές στην στους κανονισμούς, ο φόβος για τον έλεγχο, αλλά κατά την άποψή μου, ο σημαντικότερος, είναι αυτός ο φόβος του λογιστικού ελέγχου και ο φόβος των συνεπειών που θα, έχει σε περίπτωση που, θα έχετε σε περίπτωση που ο λογιστικός έλεγχος βρει προβλήματα. Θεωρώ ότι η έκθεση και η παρουσίαση που ακούσαμε είναι χρήσιμες. Μας δίνουν κάποια γενικά συμπεράσματα και κάποια θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Όμως η τάση αυτή τη στιγμή είναι να απομακρυνόμαστε από μια απλό έλεγχο συμμόρφωσης και να πηγαίνουμε περισσότερο προς μια μέτρηση των επιδόσεων. Στην αξιολόγηση των προγραμμάτων δηλαδή. Και Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα και στην Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη και στην Επιτροπή Προπολογισμού και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική τη συμμόρφωση και να πάμε προ την μέτρηση τη αποτελεσματικότητα των ελοποίηση των προγραμμάτων. Όταν μετρούμε επίδοση και αποτελέσματα, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πάψουν οι διαχειριστικέ αρχέ, οι περιφέρειε ή τα κρατημέλη να φοβούνται τον έλεγχο Μια ιδέα που θα μπορούσε να μας βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτό που ανέφερε και ο Βίκτορ για τον μοναδικό έλεγχο. Για έναν και μοναδικό έλεγχο ένα πρόγραμμα. Και συμβάσεις που να υπογράφονται ε, ε, ε, καλή την πίστη όταν γνωρίζουμε από τη μια διαχειριστική αρχή ένας φορέας διαχείρισης έχει αποδεδειγμένα ε, ιστορικό ορθής διαχείρισης, χρηστής διαχείρισης έτσι ώστε να μειώσουμε, όλα αυτά τα μέτρα είναι για να μειώσουμε τον φόβο που υπάρχει ε, του διαχειριστικού ελέγχου, τον υπερβολικό φόβο. Στα Focus Group που μας παρουσίασε ο μιλητής, μας είπε ότι άκουσε προτάσεις από, μάλλον παρατηρήσεις από εκπροσώπους των περιφερειών που μας είπαν ότι ε, το Α ή το Β δεν θα ήθελαν να το κάνουν, αλλά το κάνουν εξαιτία του φόβου του ελέγχου. Κύριος Βίτμαν. Μια και είμαι ο τελευταίος ομιλητής, δεν μένουν και πολλά να πω. Έχω καλυφθεί από όλους εκείνους που μίλησαν πριν από μένα γιατί συμφωνώ μαζί τους. Ε, το πρόβλημα όμως είναι ότι όλοι γνωρίζουμε Ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι η χιλιοστή που το συζητούμε εδώ σήμερα, αλλά δεν καταφέρνουμε να φτάνουμε σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Δεν έχουμε καταφέρει να ευκολύνουμε τη ζωή των δικαιούχων ή των διαχειριστικών αρχών. Δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει το απαιτούμενο θάρρος. Δεν υπάρχει ένας που να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να ε, επιφέρει αυτές τις αλλαγές παρά το γεγονό ότι πολλοί σε διάφορα κράτη-μέλη ε, ζητούν αλλαγές. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνη που ανέφερε ο μιλητής στο παράδειγμά του από τη Σουηδία είναι κατά την άποψή μου το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και, είναι, και, και, και, και πού είναι αυτό το πρόβλημα που εντοπίζεται, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη, μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης, στα κράτη-μέλη και στα πιο χαμηλά επίπεδα μετά, μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του δικαιούχου. Αυτό οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο. Γιατί τελικά λειτουργεί και αντιστρόφως, ο ίδιος ο δικαιούχος γίνεται επιφυλακτικός και χάνει την εμπιστοσύνη του έναντι των αρχών που θα τον ελέγξουν και ούτω καθεξής. Γι' αυτό πιστεύω ότι εξαιτία όλων αυτών στην πραγματικότητα χάνουμε τον βασικό στόχο της πολιτικής συνοχής. Γιατί, γιατί δημιουργήσαμε την πολιτική συνοχής εξ αρχής για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών της Ευρώπης συνολικά. Και χάνουμε χρόνο και σπαταλάμε πόρους σε ελέγχους και περισσότερους ελέγχους που δημιουργούν φόβο. Φόβο που παραλύει τους πάντες. Ένας λόγος που δημιουργείται αυτός ο φόβος επίσης είναι επειδή αυτοί οι έλεγχοι γίνονται με τρόπο μηχανικό δεν κάνουν διάκριση οι ελεγκτές ανάμεσα στην περίπτωση ενός αθώου και τυχαίου λάθους αφενός και περιπτώσεων διαφθοράς αφιτέρου. Τέτοιου τύπου φόβος υπάρχει και στους ίδιους τους ελεγκτές γιατί και εκείνοι ελέγχονται από μια ανώτερη αρχή και εκείνοι φοβούνται μη τους πήκανες ότι δεν έκαναν καλά τον έλεγχο. Έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Αλλά για ένα πράγμα είμαι σίγουρος, για την ε, καλή πίστη και θέληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν την δαιμονοποιώ. Ε, άκουσα και τη συζήτηση που είχαμε το πρωί εδώ στην Επιτροπή για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 ε, εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα πηγάζει από τα κράτη-μέλη και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι στο επίπεδο των κρατών μελών υπάρχουν οι διάφοροι γραφειοκράτε οι οποίοι κρύβονται πίσω από τι στίβε των εγγράφων και των κανονισμών. Ε, και τι σημαίνει κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, εξαιτία του ενό ε, προβλήματο, του ενό αθώου λάθου, δημιουργούμε ακόμα ένα μάνιο, αλλά ακόμα ένα εγχειρίδιο με νέου κανονισμού. Είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση της απάτης. Βεβαίω πρέπει να καταπολεμούμε την απάτη. Αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι όταν κάποιο ξεκινάει να σχεδιάζει ένα πρόγραμμα και του επιβάλλονται μακροσκελέστατοι κανονισμοί χιλιάδων σελίδων, πιο εύκολο είναι να κάνει και μια απάτη παρά να ακολουθήσει τους κανόνες. Γιατί ακριβώ όταν το οποίο είναι συγκεχημένο μπορεί κανείς να κρυφτεί όταν σκοπεύει να κάνει κάτι παράνομο. Είναι απλό. Φανταστείτε ότι ο κανονισμός για την υλοποίηση ενός προγράμματος είναι μόνο 50 σελίδες. Δεν θα ήταν πολύ λιγότερα τα λάθη γιατί θα, και δεν θα ήταν ταυτόχρονα και πολύ λιγότερες οι περιπτώσεις της απάτης γιατί εκείνοι που θα είχαν το, ε, τον δόλο, την, την διάθεση να ε, στήσουν μια απάτη θα γνωρίζουν ότι θα είναι εύκολο να ελεγχθούν εξαιτία αυτών των 50 σελίδων και θα τους πιάσουμε. Ενώ αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους τεράστιους κανονισμούς, με των χιλιάδων σελίδων, είναι ότι και οι έντιμοι δικαιούχοι φοβούνται και εκείνοι που θέλουν να εξαπατήσουν τα καταφέρνουν μια χαρά. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για αυτές τις παρατηρήσεις και πριν να δώσω τον λόγο στον ε, ομιλητή μας ε, για τη δευτερολογία του θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με το ρόλο μας ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως συνομοθέτες πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνε μας και να κάνουμε και εμείς αυτό που μας αναλογεί για να εξαλείψουμε τον κανονιστικό υπερθεματισμό. Αντιθέτως όμως, τι κάνουμε στην πράξη? Πολύ συχνά το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έρχεται και επιμένοντας σε λεπτομέρειες περιπλέκει το κείμενο των διαφορών κανονισμών. πολύ συχνά δεν ασχολούμαστε με το δάσος και κοιτούμε το δέντρο. Και άσκοπα περιπλέκουμε τα νομοθετήματα. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να τηρούμε τους, αυτό που λέμε, ότι θέλουμε μεγαλύτερη απλοποίηση και στις δικές μας προτάσεις και στη δική μας ε, δραστηριότητα. Δεύτερο θέμα. Κατά την άποψή μου, υπάρχει μια θεμελιώδης αντίθεση εδώ. Τι συνέβη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η Ευρώπη που ήταν κατά βάση ε, φιλελεύθερη, μεταξελίχθηκε, αλλάχθηκε σε ένα γραφειοκρατικό κτέρας. Νομίζω ότι εδώ η εξήγηση βρίσκεται στην έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης των κρατών μελών, των διαχειριστικών αρχών, των περιφερειακών αρχών και των δικαιούχων και αντιστρόφων. Και όσο λιγότερο υπάρχει εμπιστοσύνη, τόσο αυξάνονται οι έλεγχοι. Τρίτη παρατήρηση. Είναι κάτι για το οποίο προσωπικά τουλάχιστον είμαι πεπισμένος. συχνά έχουμε την τάση όταν υπάρχει έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης προσπαθούμε να την καλύψουμε και να την αντικαταστήσουμε υπερβάλλοντας στους ελέγχους και στην τιμωρία. Και αν συνεχίσουν οι πολίτες μας, αν συνεχίσουν οι λαοί της Ευρώπης να προσλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν οργανισμό που έρχεται να ελέγχει και να τιμωρεί, Πιστεύω ότι η έλλειψη εμπιστοσύνη και η καταδίκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση από του Ευρωπαίου πολίτε θα αυξάνει όλο και περισσότερο. Ε, προσπάθησα να συνοψίσω τη συζήτηση, θα δώσω το λόγο και στην εκπρόσωπο τη Επιτροπή, τη ομάδα μελετών. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά των ομιλητών για να μην ξεχάσω κανέναν. Ο πρώτος ομιλητής ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία διαδικασία για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό κυριαρχεί πολύ στη συζήτηση. Αλλά το ερώτημα είναι το εξή. Υπάρχουν διάφορα διοικητικά συστήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργούσε ένα ενιαίο σύστημα. Και είναι και διαφορετικέ οι κουλτούρες, οι νοοτροπίε, οι διοικητικοί πολιτισμοί κάθε κράτο Δεν είναι τόσο εύκολο να είναι ενιαίες οι διαδικασίες. Υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμών και χειρισμών, αλλά ε, πρέπει να ξέρουμε ότι διαφέρουν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους και οι περιφέρειες πόσο μάλλον. Δεύτερος ο μιλητής από την Τσεχική Δημοκρατία ρώτησε για τη συμμετοχή μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων ή νομικών οργανώσεων αρκετά νωρίς έτσι ώστε να ελέγχουν ε, την ε, νομοθεσία στο νομοπαρασκευαστικό στάδιο. Μα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα βοηθούσε πάρα πολύ η εκ των προτέρων συνεννόηση και ακριβώ δεν δημιουργούνται και αδικαιολόγητοι φόβοι λόγω παρεξηγήσεων ή παρανοήσεων. Ε, ένα είδος αντικτή που θα μπορούσε να λειτουργεί στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά ε, πολλέ ε, πολλές φορές ο υπερθεματισμός ε, έρχεται στο στάδιο της ερμηνείας των διαφόρων προγραμμάτων και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εκ των προτέρων. Δηλαδή εδώ υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ε, στα εργαλεία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ο συνάδελφος, ε, ο μιλητής μάλλον από τη Σουηδία, ανέφερε το φόβο των ελεγκτών και το ρόλο τους. Μα δεν φοβούνται τους ίδιους τους ελεγκτές φοβούνται τον έλεγχο. Ε, ακριβώς είναι ο φόβος του επιθεωρητή. Πώς θα το διαβάσει, πώς θα το ερμηνεύσει, πώς θα το πάρει. Ε, δηλαδή πολλές φορές δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο κόσμος φοβάται τόσο πολύ τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται τόσος φόβος. Και έχουμε την αίσθηση καμιά φορά στις ότι πρέπει να το λέμε. Ε, ένας ε, διάλογος νωρίς μεταξύ των επιθεωρητών και εκείνων που εφαρμόζουν το πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Αν έρθει ο ελεκτή και πει ότι κοιτάξτε, εμεί το βλέπουμε έτσι και το ελέγχουμε έτσι και ψάχνουμε αυτό, τότε θα ξέρει πού βαδίζει ο δικαιούχο και θα υπάρχει διάλογο και διαφάνεια που θα βοηθούσε πάρα πολύ. Αυτή η ιδέα για τι πλατφόρμε για τους πολύ μικρούς ε, δικαιούχους όπου είναι πολύ βαριές οι διαδικασίες και πολύ περίπλοκες και δεν τολμούν μόνοι τους να ε, κάνουν αυτό το βήμα. Θα λειτουργούσε αυτή η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και μια έτσι, επίκριση που εκφράζεται εκεί, γιατί δεν είναι δωρεάν. Ε, Υπήρχε ένα συγκεκριμένο κόστος ε, των δημιουργών αυτής της πλατφόρμας που παίρνουν πολλά χρήματα ε, ω μεσάζοντες ας πούμε. Εμείς θέλουμε τα λεφτά να πηγαίνουν στους τελικού δικαιούχου και όχι σε διάφορους μεσολαβητές, έστω και αν είναι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και αν βοηθούν ε, τους μικρούς να συμμετέχουν. Τι άλλο. Συνάδελφοι από τη Ρουμανία για την περιπλοκότητα και την εναρμόνιση. Το πρόβλημα ποιο είναι. Οι ελεγκτές δεν ελέγχουν μόνο την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και την εθνική. Ξέρω μια περίπτωση στη Σουηδία που έλεγξαν την ευρωπαϊκή συμμόρφωση ε, ε και εκεί ε, ε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά γνώρισαν τη Σουηδική που ήταν αυστηρότερη. Οπότε πρέπει πάντα να σεβόμαστε το κάθε νομικό πλαίσιο και θεσμικό. Δεν μπορούμε λοιπόν να εναρμονίσουμε, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα πλαίσια. Λοιπόν, για τους ελέγχους Δεν είναι τόσο εύκολο να εναρμονιστούν, να γίνουν ενιαίοι. Έγιναν πολλές ερωτήσεις για συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν κατάφερα να σας αναφέρω μερικά, ε, γιατί θα ξεπερνούσε κατά πολύ το χρόνο μου. Στην έκθεση όμως θα βρείτε διάφορα παραδείγματα για ποιους λόγους γίνεται αυτός ο υπερθεματισμός και περιγράφουμε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου μπορείτε να ανατρέξετε. Είπατε να φύγουμε από την συμμόρφωση και να πάμε στις επιδόσεις. Η έλεγχη μπορούν να γίνουν στις επιδόσεις και όχι στη συμμόρφωση, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή εκεί. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς δείκτες και ξεκάθαρα συστήματα. Γιατί υπάρχουν διάφορα επίπεδα ελέγχων και δεν είναι πάντα ξεκάθαρες οι λεπτομέρειες. και καλό θα ήταν ε, σε πολύ πρώιμα στάδια να γίνονται οι συνεννοήσεις για να απλουστεύονται τα πράγματα. Έγινε και μια ερώτηση για το πώς θα μπορούσε να διευκολυνθεί η κατάσταση. Σας το είπα και προηγουμένως. Ένα από τα παραδείγματα ε, ε, και αυτά που μας ζητούν οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι είναι να υπάρχει νωρί συνεννόηση μεταξύ των ελεγκτών και των ε, φορέων για να ξέρουν ε, τι τους ζητούν πριν την εκτέλεση του προγράμματος. Έτσι θα δημιουργηθεί και μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων ενεχομένων, των ελεκτών, των δικαιούχων, των αρχών αυτοδιοίκησης για να σπάσει αυτή η ατμόσφαιρα φόβου που κάνει τους ανθρώπους να είναι υπερβολικά επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Και αυτό με φέρνει σε αυτό που είπε ο πρόεδρος. Να δημιουργηθεί μια εμπιστοσύνη, να ξέρουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε και να μην έχουμε τη φοβέρα κάθε φορά ε, του ελέγχου, του, των υπερβολικών μέτρων, της εμπιστοσύνης και της δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπόμα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την ε, Μονάδα Μελετών ε, το τμήμα Β για την ε, ε, συμβολή τους σε αυτές τις εργασίες. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας. Ξέρετε ότι στις 23 ε, Ιανουαρίου που μας πέρασε εξετάσαμε για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων την έκθεση πρωτοβουλίας του συναδέλφου Μπούντα που στόχο έχει να ενισχύσει τη συμμετοχή των εταίρων και τη διαφάνεια των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διευθυντικών και Επενδυτικών Ταμείων. Διατυπώσατε διάφορες προτάσεις. Θα σας δώσω το λόγο και να θυμίσω μόνο ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 3η 28 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Ο εισηγητής έχει το λόγο και μετά θα ακούσουμε τους διάφορους κοιόδες εισηγητές. Uh, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάμπερτ για την υποστήριξή του στη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της έκθεσης, καθώς και τους συντονιστές. Διότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας ήταν απαραίτητη για να αυξηθεί η ορατότητα της πολιτικής ε, ε, συνοχής. Αυτό είναι ένα βασικό ε, μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του οποίου μειώνονται οι διαφορές ανάμεσα στις περιφέρειες, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η απασχόληση και στηρίζεται η ανταγωνιστικότητα στις διάφορες περιφέρειες της Ένωσης. Οι επενδύσεις ε, που γίνονται από την ε, πολιτική συνοχή έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία των κρατών μελών, πράγμα που έχει συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά που δυστυχώς τα πλονεκτήματα που απορρέουν από αυτές τις επενδύσεις δεν γίνονται πάντοτε αισθητά όπως θα θέλαμε από πλευράς των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή την, σε αυτή την έκθεση ξεκινήσαμε από το γεγονό ότι η πολιτική συνοχή χρηματοδοτείται από ένα προπολογισμό 800 60 εκατομμύριων ευρώ, αλλά ο συντονισμός δεν ήταν πάντοτε πιο αποτελεσματικό. Και όπως λέω και στην εκθεσή μου, μόνο το 1 τρίτο των ερωτηθέντων από το Ευρωβαρόμετρο του 2015 έχουν, είχαν ακούσει να γίνεται λόγος για έργα που συγχρηματοδοτούνται από, την πολιτική, από το κονδύλιο της πολιτικής συνοχής ε, και που βελτίωσαν την καθημερινότητά τους. Μόνο το 1 τρίτο των ερωτηθέντων γνώριζαν την ύπαρξη αυτής της πολιτικής αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα κλίμα δυσπιστίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ε, ε, ανάπτυξης των συστημάτων, ε, μάλλον των ακραίων κομμάτων, του Brexit, μας κάνουν όλα αυτά, να κάνουν μάλλον τον κόσμο να αμφιβάλλει, όπως και οι διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης. Η έλλειψη επικοινωνίας έχει συμβάλει σε αυτήν την στη δημιουργία αυτού του κλίματος. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για το μέλλον, γιατί όπως είπαμε βάσει τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο το 7% των ανθρώπων που ρωτήθηκαν γνώριζαν ότι γίνονται επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο άλλο άκρο ήταν η Πολωνία όπου το 73% των ερωτηθέντων γνώριζαν το θετικό αντίκτυπο των project της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή όπου ζουν ε, τεράστια διαφορά ανάμεσα στο 7% της Βρετανίας και το 73% της Πολωνίας. Το πρώτο συμπέρασμα που μπορούμε να ανασύρουμε είναι ότι χρειάζεται καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στις δημόσιες αρχές, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους αλλά και την κοινωνία των πολιτών έτσι να, να γνωστοποιούνται καλύτερα οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αυξάνεται το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών για αυτήν. Η πρωτοβουλία λοιπόν δομείται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο, η έκθεση μάλλον πρωτοβουλία δομείται σε τέσσερα κεφάλαια. Πρώτα έχουμε τι γενικέ παρατηρήσει, όπου γίνεται μια ανάλυση τη ισχύουσα κατάσταση ω σημείο εκκίνηση, ώστε να υπάρξει επικοινωνία για τα αποτελέσματα της, της πολιτικής συνοχής και το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και αναφέρει επίσης τους περιορισμούς που εξακολουθούν να υφίστανται για μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία στο τρίτο τμήμα γίνεται λόγος για συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της επικοινωνίας και την ε, εμπλοκή των εταιρών στο δεύτερο ήμιση της χρηματοδοτικής περίοδου 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόταση κανονισμού Omnibus. Εδώ προσπάθησα να περιλάβω απτούς στόχους, εφικτούς μάλλον στόχους. Στο τέταρτο δε κεφάλαιο εστιάζω στα μέτρα προώθησης της επικοινωνίας, κυρίως στην ανάγκη να συμμετέχουν οι εταίροι και οι πολίτες στην προοπτική μετά το 2020, γιατί ε, θα πρέπει να εστιάσουμε και, για, ε, και στο ε, μετά το 2020 εποχή. Χρειάζονται δηλαδή και νέα μέσα επικοινωνίας, αλλά και εντοπισμός ενός πλαισίου, μέσα στο οποίο οι ίδιοι δικαιούχοι θα απειχούν ε, το όφελος ε, που έχουν αποκομίσει από τα κονδύλια της συνοχής. Χρειάζονται δηλαδή δείκτες που να μετρούν την αποτελεσματικότητα των ε, μηνυμάτων ορατότητα όσον αφορά την πολιτική συνοχής και είναι ευθύνη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, γιατί αυτές είναι οι αρχές οι οποίες ε, έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες. Οι τοπικές αρχές χαίρουν ψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνη από πλευρά των πολιτών, γιατί ακριβώς έρχονται σε επαφή μαζί τους. Είναι σημαντικό αυτό για να βελτιωθεί η επικοινωνία. Και επίσης είναι απαραίτητο το μήνυμα αυτό να λαμβάνει υπόψη και τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα του δικαιούχου. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε ποιες πρόοδοι έχουν σημειωθεί σε θέματα επικοινωνίας που διαφέρουν από μια περιφέρεια στην άλλη. Η δε τεχνική αρρωγή που συνδέεται με το Ταμείο Εύση θα πρέπει να προβλέπουν μεγαλύτερο μερίδιο για την επικοινωνία ε, γιατί η επικοινωνία αυτή τη στιγμή περιλαμβάνεται αλλά σε πολύ χαμηλό ποσοστό στο πλαίσιο της τεχνικής αρρωγής. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν δύο συνιστώσεις. Η μία να στα, ίδια τα προγράμματα και ένα άλλο τμήμα να αφιερώνεται στην ε, υλοποίηση αυτών. Η συμμετοχή των εταίρων είναι δύσκολη ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε οι εταιρικέ αυτές σχέσεις να αγκαιώνται μεγαλύτερη συμμετοχή και να δίνουν περισσότερη ευθύνη για την υλοποίηση τα δε αποτελέσματα του Ταμείου Συνοχής δεν είναι άμεσα ορατά όπως ε, αυτά του ΕΦΣΥ. Γι' αυτό και η στρατηγική επικοινωνία στο ΕΦΣΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει μια δεφική πτυχή. Ο Επίτροπος Κατάινεν είπε χτες ότι υπάρχουν μέλη τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα του προγράμματος Juncker και εκπρόσωποι των σημαντικών ε, μάλιστα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των κρατών υποστηρίζουν ότι ποτέ δεν άκουσαν, δεν έχουν ακούσει καν για την ύπαρξη των δυνατοτήτων χρηματοδότησης από το σχέδιο Juncker. Πρέπει λοιπόν να βρούμε και να υιοθετήσουμε μέτρα που θα σχετίζονται με, ε, που θα υποχρεώνουν στην ε, επικοινωνία όσον αφορά τα project που χρηματοδοτούνται από το ΕΦΣΙ και από το Ταμείο της Συνοχής, έπειτα μεγαλύτερο συντονισμός, αλλά και αυτό να γίνεται μέσα από τις αρχές διαχείρισης και από τους ίδιους του δικαιούχους. Και έπειτα, μιλώντας για διοικητικές διαδικασίες, θα είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και εδώ θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι οι πρόοδοι είναι πολύ διαφορετικές στα διάφορα κράτη-μέλη και σε αυτό το πλαίσιο εμείς είμαστε υπέρ μέτρων που προβλέπουν διαδικασίες ομοιόμορφες, τουλάχιστον για ορισμένε επιτυχίες σε επίπεδο κρατών μελών. Η εναρμόνιση ε, των αποτελεσμάτων της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο της επόμενης στρατηγικής επικοινωνίας, δηλαδή επικοινωνία προς τα έξω όσον αφορά τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής, όπου η Κομισιόν θα πρέπει να υιοθετήσει διάφορες στρατηγικές επικοινωνίες ε, και για τα κράτη που είναι καθαροί εισφορείς και για εκείνα που είναι καθαροί δικαιούχοι δύο διαφορετικά επίπεδα επικοινωνίας και παραθέτω ένα παράδειγμα. Αν ε, μία επιχείρηση ενός κράτους που είναι καθαρός ε, ε, εισφορείς ε, θα πρέπει να μπορεί να δείξει ότι και αυτή η επιχείρηση κερδίζει, κερδίζει καθώς αυξάνεται το ΑΕΠ της εν λόγω χώρας. Οπότε οι πολίτες της χώρας που είναι καθαρός εισφορέας να γνωρίζουν ότι ωφελούνται και αυτοί από τα κονδύλια των διορθωτικών ταμείων μακροπρόθεσμα μόνο με τη συμμετοχή όλων των εταίρων ε, θα μπορέσουν να ωφεληθούν κιόλας όλοι. Μεγα, περισσότερη πολιτική ευθύνη, να αναπτυχθούν δηλαδή πλατφόρμες μέσα με βάση τα σημερινά μοντέλα συμμετοχή διακυβέρνησης και με τη συμμετοχή και την ανάμεξη των ίδιων των πολιτών. Μια συμμετοχική διαδικασία για τον καθορισμό των ε, κονδυλίων και των ταμείων, που θα μπορούν δηλαδή οι πολίτες να σχηματίσουν και να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητες τους όσον αφορά τις επενδύσεις στην περιοχή τους. Και έτσι ο πολίτης θα αισθάνεται μέρος όλης αυτής της διαδικασίας και θα φέρει και ευθύνη όσον αφορά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και αυτό φυσικά θα αυξήσει και την ε, ορατότητα. Ευχαριστώ λοιπόν όσους συνεργάστηκαν για αυτή την έκθεση. Να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Τόγιαν και τον κύριο που είναι ε, ε, από τη γραμματεία του ΕΛΚ, την, τον κύριο Στόνα από την Επιτροπή μας και επίσης ευχαριστώ για τη στενή συνεργασία στην Επιτροπή των Περιφερειών. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Κύριε συνάδελφοι, θα δώσω τώρα το λόγο στους ασκηώδεις συζητητές. Mm Ζουφρίντα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ ε, και ευχαριστώ τον κύριο Μπούντα για αυτή την έκθεση που περιλαμβάνει τα κεντρικά στοιχεία που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ επανειλημμένα σε αυτήν την Επιτροπή. Στην τελευταία μας επαφή με την Επίτροπο Κρέτσου εστιάσαμε την προσοχή στα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής και κυρίως στο πώς μπορούμε να διαδώσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Δύο επίπεδα, ένα γενικότερο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα άλλο πιο ιδιαίτερο για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Αυτό που αφορά το μέλλον της Ένωσης μας οδηγεί να διαπιστώσουμε την ε, απομάκρυνση και την δυσπιστία των πολιτών προς την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι πολύ σοβαρό που οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν καταλαβαίνουν και δεν γνωρίζουν πώς παρεμβαίνει η Ευρώπη στην ανοικοδόμηση δρόμων, στην, στο ευρυζωνικό ίντερνετ κτλ. Έπειτα ε, η, το, η πολιτική συνοχή στην ουσία δέχεται επιθέσεις από το εσωτερικό και πρέπει να αντιμετωπίσει, είναι μια σημαντική μάλλον γραμμή του προπολογισμού και τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα ικανοποιητικά και κυρίως δεν είναι πάντα ορατά. Και για να μπορέσουμε να αντιπαράσουμε αυτές τις δύο δυνάμεις που θέλουν να ε, απαξιώσουν την ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να τονίσουμε εμείς τα αποτελέσματα και τις επιτυχίες μέσω ε, των, ε, τα όσα πετυχαίνουμε μέσω αυτών των ταμείων, των διευθυντικών και των επενδυτικών δεν είναι ε, κόλπο, είναι πραγματικότητα και αυτό σημαίνει συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων πρώτα και μετά στην διαδικασία αξιολόγησης στην συνέχεια. Ο συνάδελφος υπογραμμίζει στην εκθεσή του ότι η ορατότητα τη πολιτική συνοχή βασικά είναι θέμα των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Εγώ πιστεύω πως είναι και μια γενικότερη στρατηγική που θα πρέπει να οικοδομηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει στοχευμένη δράση με δύο στόχους. Ο πρώτος να καλυφθούν ε, οι προκαταλήψει όσον αφορά την ανεπάρκεια και την ε, αδυναμία των διευθυντικών ταμείων. Και ένα δεύτερος άξονας θα πρέπει να είναι ε, αυτός που ορίζει και καθορίζει, δείχνει πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βοηθά στην ανάπτυξη των διαφόρων ε, περιφερειών. Γι' αυτό θα μπορούσε η Επιτροπή, οι περιφέρειες και οι αρχές Διαχείριση σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να δουν πώς, ποιο είναι το καλύτερο μέσο ενημέρωσης. Γιατί δεν αρκεί πλέον όπως κάποτε να βάζουμε την πλακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, πινακίδα του έργου. Χρειάζονται περισσότερα μέσα. Πρέπει κατά τη γνώμη μου να ανακοινώνονται και να υπάρχει επικοινωνία για όλες τις φάσεις ε, που πολλές φορές άλλωστε τα έργα αυτά κρατάνε χρόνια και χρόνια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είναι φωτισμένες όλες οι φάσεις όχι μόνο ανακοινώσεις ε, στην έναρξη ενός ε, έργου, γιατί αυτό μετά μπορεί να έχει και καταστροφικό εφέ στην ε, κοινή ε, νου, αν δεν μπορούμε τελικά να, να δει ο κόσμος τα διάφορα βήματα ολοκλήρωση του ίδιου του project. Γιατί το κενό καλύπτεται από τους λαϊκιστές, αυτό συμβαίνει πολύ συχνά με πληροφορίες οι οποίες είναι λάθος, απλουστευτικές, και παραπλανητικές. Να σας πω τέλος ότι οι τροπολογίες που θα υποβάλω θα στόχο έχουν περισσότερο να προωθηθεί η σωστή ορατότητα των επιτυχιών της πολιτικής συνοχής και στα διάφορα βήματα υλοποίηση των project. Συμφωνώ με τον εισηγητή για το γεγονό ότι η τεχνική αρρωγή θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα κονδύλι ειδικά για την ε, επικοινωνία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει και κατευθυντήριες γραμμές, μια πλατφόρμα να οργανώσει βραβεία, ας πούμε, για το πώς, επίσης, γραφεία που θα βοηθάνε στο πώς οργανώνεται ένα site ε, στο ίντερνετ, να υπάρχει ένα κοινός ε, ηρμός, ε, ε, και επίση η Κομισιόν θα πρέπει να ετοιμάσει μια βάση δεδομένων που θα είναι εύκολα προσιτή και που θα περιλαμβάνονται όλα τα, τρέχοντα ε, project και το στάδιο πρόοδου τους με φωτογραφίες πριν και μετά. Αυτό κάνουν και τα ιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικέ υπηρεσίες, γιατί να μην το προωθήσουμε άμεσα. Ε, επίσης, επαφή με τα τοπικά μέσα ενημέρωση πρέπει να υπάρχει να δίνεται αναφορά για όλες τις φάσεις των έργων, να ε, διηγούνται δηλαδή ιστορίες. Και επίσης θα πρέπει να διασπιστεί και ένα βραβείο για το καλύτερο project που έχει υλοποιηθεί κάθε χρόνο. Ναι, ναι, κλείνω. Και λέω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε ένα ακαδημαϊκό στυλ, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, να μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε τα όσα έχουν γίνει, να συγκριθούμε με τις υπόλοιπες περιφέρειες στην Ευρώπη. Και γι' αυτό θα πρέπει να δράσουμε και με την αξιολόγηση των πεπραγμένων από τις τοπικές αρχές και βέβαια θα πρέπει αυτή την απόφαση και την κρίση να την κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την e η κυρία Τόμασετς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπούντα για το σχέδιο έκθεσής του. Γενικά υποστηρίζω τα περισσότερα σημεία και τις προτάσεις του. Είναι πάρα πολύ σωστό ότι είναι διαφορετική συνειδητοποίηση ε, από χώρα σε χώρα για τα αποτελέσματα της πολιτικής των διαθωτικών ταμείων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη επικοινωνία για να προβάλλουμε τα θετικά στοιχεία και το θετικό αντίκτυπο και την ευεργετική επίδραση που έχουν τα διαθωτικά ταμεία και στη ζωή των πολιτών και στην οικονομία. Και να κάνουμε και μία σύγκριση, ε, ε όχι όμως μεταξύ του ΕΦΣΙ και των διαθωτικών ταμείων, ε, δεν υπάρχουν στοιχεία που να λένε ότι ε, τα αποτελέσματα ε, της συνοχής είναι καλύτερα από το ΕΦΣΥ. Πολλά από τα έργα που ενισχύει το ΕΦΣΥ είναι μακράς πνοής και δεν ευσταθεί η σύγκριση. Υποστηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως και τα ταμεία της συνοχής. Ευχαριστώ. Κύριε ευχαριστώ εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Θέλουμε και εμείς να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπούντα για το σχέδιο έκθεσης. Συμφωνούμε ότι η αύξηση της προβολής και της ορατότητας και της διαφάνειας ε, των διαρθρωτικών ταμείων είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν θα πρέπει να προβάλλουμε με διαφορετικό τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διορθωτικά ταμεία. Ε, αν είναι θετική η προβολή, ο κόσμος θα αντιλαμβάνεται καλύτερα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προσπάθειές της. Θα πρέπει να βασιζόμαστε όμως στα αποτελέσματα και θα πρέπει να έχει και περιεχόμενο επικοινωνία και αντικείμενο και όχι γενικά και αόριστα. Στην Ολλανδία υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι δεν θα πρέπει να επικοινωνείς για την επικοινωνία. Πρέπει να έχεις κάτι να πεις, ένα μήνυμα. Λοιπόν, χρειάζεται πληροφορία για τις δυνατότητες χρηματοδότησης, πώς μπορεί κανείς να έχει καλύτερη πρόσβαση ένας πιθανός δικαιούχος που θέλει επιδότηση. Και από την άλλη έχουμε και την επικοινωνία για τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής προς τους πολίτες, όχι τους δικαιούχους στο γενικό κοινό. Μου λείπει λίγο στην παράγραφο 18 αυτή η διάκριση. Ο εισηγητής μιλάει για μετάφραση σε διάφορες γλώσσες. Για ποιον όμως, για τους δικαιούχους στο ΕΣΠΑ της κάθε χώρας. Εγώ δεν θέλω να δαπανίσω πολλά λεφτά εκεί στις μεταρρυθμίσεις για το προφανές. Ε, ή όταν το κοινό είναι αμυγός εθνικό, γιατί να το μεταφράσω σε όλες τις γλώσσες. Και στην παράγραφο 19, Task Force για την επικοινωνία με ε, συμμετέχοντες από διάφορα επίπεδα, αυτό θα μπορούσε να έχει νόημα, αλλά στα πλαίσια ενός ε, επιχειρησιακού προγράμματος, εθνικό επίπεδο, όχι ευρωπαϊκό, που να αφορά ένα επιχειρησιακό σχέδιο σε μια χώρα. Αντιμετωπίζω κάποιες δυσκολίες και με την παράγραφο 24 για την εισαγωγή ενός δεσμευτικού ποσοστού τεχνικής βοήθειας. Ε, που θα πρέπει να μπει στην άκρη για την επικοινωνία. Μα η τεχνική βοήθεια ε, προβλέπει ε, κονδύλια για την επικοινωνία ήδη. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τέτοια ποσοστά υποχρεωτικά. Η τεχνική βοήθεια έχει ε, σκοπό να βοηθήσει τις περιφέρειες και του οτά να εφαρμόζουν την πολιτική συνοχής. Και στην ίδια παράγραφο ζητάει ο εισηγητής υποχρεωτικά κριτήρια επιλεξιμότητας που να συνδέονται με την ποιότητα της επικοινωνίας. Και πάλι λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω. Αφετηρία της επιλογής ενός προγράμματος θα πρέπει να είναι η ποιότητα του προγράμματος και όχι της επικοινωνίας μόλις τελειώσει. Και έχω και μια ερώτηση στην παράγραφο 26. Ζητεί ο εισηγητή να συμμετέχουν οι ενεχόμενοι stakeholders στη διαδικασία κατάρτιση του προπολογισμού. Πώ ακριβώ το σκέφτεστε αυτό. πώ θα βελτιωθεί και σε ποιο επίπεδο, πού θα συμμετέχουν. Γιατί εγώ βλέπω κάποιες δυσκολίες και κάποιες εντάσεις να δημιουργούνται και τριβές κυρίως μεταξύ των διαχειριστικών αρχών που θα συμμετεχουν γιατι εγω βλεπω κάποιε δυσκολίε και κάποιε εντάσει να δημιουργουνται και τριβε κυριως μεταξυ των διαχειριστικων αρχων που δουλευουν με προκηρύξεις, με δημοπρατήσεις και με ανταγωνισμό για να βρουν το καλύτερο έργο και από την άλλη έχουμε τις επιθυμίες και τις απαιτήσει των ενδιαφερομένων να συμμετέχουν και στη διαδικασία κατάρτισης του προπολογισμού. Πώς το σκέφτεστε αυτό συγκεκριμένα στην πράξη να λειτουργεί. Πώς το έχετε φανταστεί. Και στην παράγραφο 30 επίσης κάνετε μια πρόταση που νομίζω ότι ξεφεύγει. Να δημιουργηθεί μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας. Αμφιβάλλω για την εφαρμογή. Νομίζω θα πρέπει να αποφύγουμε διπλοδουλειές και επικαλύψεις. Υπάρχει ένα πόρταλ με τα δεδομένα. Ας μην πολλαπλασιάζουμε τώρα την επικοινωνία, ε, να μην εντείνουμε προσπάθειες με επικαλύψεις και διπλές δουλειές, γιατί έχουν και κάποιο κόστος όλα αυτά τα πράγματα και είναι χρήματα των φορολογουμένων. Θα πρέπει να πιάνουν ε, τόπο με τρόπο και όχι όπως να είναι. Και επίση κάπω θα πρέπει να συνδέσουμε την έκθεση αυτή με το ρόλο των Εθνικών Γραφείων Επικοινωνίας και Ενημέρωση. Υπάρχουν ένα σωρό δίκτυα εκεί σε όλα τα κράτη-μέλη, ε, συμμετέχουν σε δραστηριότητε, πολύ ενημερωτικές και επικοινωνίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει ε, τη δικτύωση, την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων αυτών και καλό θα ήταν να το γράψουμε και στην έκθεσή μας. Θα κάνω κάποιες τροπολογίες και προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις, του υπολείπους, για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η τόσο σημαντική αυτή έκθεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ τον συνάδελφο για αυτή την έκθεση. Είναι ένα σχέδιο έκθεση που περιλαμβάνει διάφορα ενδιαφέροντα σημεία και όλα έχουν, ε, τονίζουν, όχι, μάλλον εμπίπτουν όχι μόνο στην πολιτική συνοχή, αλλά και στη σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες, ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους πολίτες. Και ξεκινώ από κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Δεν μπορούμε παρά να δεχτούμε όλες τις πρωτοβουλίε που δίνουν σωστό, ε, σωστή έμφαση στην πολιτική συνοχή και δεν, ε, χωρίς να σημαίνουν περαιτέρω δαπάνε να σε σχέση με τον προπολογισμό. Από την πρακτική άποψη είμαστε υπέρ οποιασδήποτε ανταλλαγή καλών πρακτικών. Ωστόσο, θεωρούμε πω είναι απαραίτητο για να υπάρξει σε πραγματική αξιοπιστία τη πολιτική συνοχή να τονίσουμε τόσο τι καλέ όσο και τι κακέ πρακτικέ μέσω ε, βάσεων δεδομένων ναι, που όμως να μην περιορίζονται σε μια περιγραφή του project και των ε, δαπανών, αλλά που ε, επιτρέπουν στους πολίτες να επαληθεύσουν τόσο την προσθέμενη αξία όσο και την αξία των περισσότερων project που έχουν υλοποιηθεί και κατά πόσο είναι χρήσιμα ή όχι σε σχέση με κάποια ε, συγκεκριμένη περιοχή. Και εκεί δηλαδή μέγιστη διαφάνεια. Πολλέ φορέ οι ίδιε οι εθνικές αρχές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εκλογικέ αναμετρήσει, ε, παρουσιάζουν την πολιτική συνοχή ως ένα αποδιοπομπαίο τράγο ε, για τις δίθεν δαπάνε και σπατάλες των Βρυξελών. Είμαστε λοιπόν ε, κάθε φορά έχουμε πρόβλημα όσον αφορά το προγραμματισμό 2007-2013, ε, την καθυστερημένη έναρξη των προγραμμάτων της περίοδου 2014 με 2020 και την περίοδο μετά το 2020. Η τοπική λοιπόν και περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι πολύ σημαντική δεν μπορούμε, πα, μάλλον όλα αυτά τροφοδοτούν την προπαγάνδα κατά ε, υπέρ μάλλον του ευρωσκεπτικισμού. Από την έναρξη, τη, το σχηματισμό των, του κόμματος των πέντε αστέρων έχει καθορίσει μια αντιευρωπαϊκή πολιτική. Ε, ε, ε, θεωρούμε πως δεν θα πρέπει να ξεκινήσει η καταστροφή λόγω μηδενιστικών σλόγγαν, ξενοφοβικών σλόγγαν που θυμίζουν φαντάσματα του παρελθόντος. Εμείς είμαστε σε ένα τρίτο δρόμο επικριτικό αλλά επικοδομητικό με προτάσεις συγκεκριμένες και ακριβείς για όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Στην πολιτική συνοχή συγκεκριμένα κάνω την εξή ερώτηση στους συναδέλφους σήμερα που είναι εδώ και που αντιστάθηκαν σε αυτή τη μακριά μέρα εργασίας για τρία θέματα πολύ καυτά και επίκαιρα. Άρθρο 23 για την ε, μακρο ε, την οικονομική την συμπερίληψη της χρηματοδότησης των project που να υπολογίζονται στην ε, μείωση του χρέους. Αυτά όλα δεν συμβάλλουν στον ευρωσκεπτικισμό. Η συμμετοχική διακυβέρνηση που ανέφερε ο συνάδελφος νομίζω πως ε, ναι, σημαίνει πιο ε, συμμετοχική διαδικασία σε αυτή την προσπάθεια συνεργασίας. Ευχαριστώ. Δύο λόγια τώρα η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση. Θεωρούμε ότι περιλαμβάνει χρήσιμες συστάσεις και προτάσεις και εμείς κατευθυνόμαστε, εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση να βελτιώσουμε την προβολή και τη δημοσιότητα της ε, πολιτικής συνοχής έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν τι ωφέλη αποκομίζουν από τις περιφερειακές πολιτικές. Υπάρχουν όμως χώρες, ιδίω εκείνε που έχουν ιδιαίτερα ε, ευεργετηθεί από τα περιφερειακά προγράμματα, αναφέρεται την Πολωνία, μπορούμε να μιλήσουμε για την, Πολωνία, ε, συγγνώμη, για την Ουγγαρία επίσης και τι Βαλτικέ χώρες, όπου τα πράγματα είναι καλύτερα, όπου οι πολίτες γνωρίζουν. σε ποσοστά άνω του 80%. Και το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι από αυτούς τους πολίτες που δηλώνουν ότι γνωρίζουν, ε, έχουν, τα τρία τέταρτα έχουν και μια θετική γνώμη για τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών. Αναφέρθηκε το δίκτυο των ε, συναδέλφων που ασχολούνται με θέματα ε, επικοινωνίας. Συνεργαζόμαστε τακτικά με αυτούς και προσπαθούμε να μοιραζόμαστε βέλτιστες πρακτικές Γίνονται δύο ή τρεις ε, συναντήσεις κάθε χρόνο και ε, μοιραζόμαστε μεταξύ μας τις καλύτερες ιδέες. Επίσης προσπαθούμε να παράσχουμε εκπαίδευση, εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα όπως είναι οι τεχνικές επικοινωνίας. Και σκοπεύουμε να εντείνουμε αυτή την προσπάθεια. Τέλος. Μιας και αναφέρθηκε το ζήτημα της προκήρυξης που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα σχέδιο δράση, μάλλον η έκκληση που απευθύνθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει ένα σχέδιο δράσης. Ε, το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι εργαζόμαστε για να το προετοιμάσουμε ε, και εμείς προσπαθούμε κατά τη διάρκεια του 2017 την πλευρά της Επιτροπής να αυξήσουμε τις προσπάθειες μας για περισσότερη δημοσιότητα, για περισσότερη προβολή. Και ευχαρίστω να συνεργαστούμε μαζί. Ευχαριστώ, δίνω το λόγο στον εισηγητή. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ε, σε όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμα ε, αυτά που είπαν. Είναι όντως σημαντική η έκθεση. Όχι επειδή είναι δική μου. Και είπε η κυρία Τζουφρίντα ότι είναι κρίμα που ε, συμβαίνουν τόσα πολλά, τόσα θετικά και καλά στην Ευρώπη και ο κόσμος δεν τα παίρνει είδηση. Βεβαίως και είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Μετά κάποιος ρώτησε γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα ποσοστό ε, για ε, την επικοινωνία και για τη διαφήμιση γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτά που έχουμε σήμερα δεν επαρκούν. Αν θέλετε θα το συζητήσουμε. Εγώ μια πρόταση έκανα, δεν έβαλα συγκεκριμένο ποσοστό. Ε, κάθε φορά εξαρτάται από το εκάστοτε πρόγραμμα πόσο ε, σημαντικό είναι το έργο ε, όχι. Υπάρχει στον προϋπολογισμό κάθε έργου ένα ποσό για προβολή και διαφήμιση. Κάτι άλλο τώρα που ήθελα να αναφέρω έχει να κάνει με τη συμμετοχή των πολιτών σε όλες αυτές τις διαδικασίες και τα έργα που χρηματοδοτούνται και από ευρωπαϊκά κονδύλια. Εγώ κατάγομαι από μία πόλη που έχει την ευτυχία και την τύχη να έχει δήμαρχο ο οποιος τρια τρία-τέσσερα χρόνια ήταν πρωθυπουργός. Και κάθε φορά που έχει προϋπολογισμό ε, ρωτάει τους πολίτες, τους δημότες του, ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι θέλετε να κάνουμε στο Δήμο, ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα ε, για τη δημοτική πολιτική ή και για άλλες πολιτικές. Θα μπορούσε αυτό να επεκταθεί και σε άλλα επίπεδα διακυβέρνησης. Απευθύνεται στους δημότες. Ο Δήμαρχος λέει έχω τόσα λεφτά, έχω αυτούς τους στόχους από το 1 μέχρι το 10 και αποφασίζουν οι πολίτες και λένε τη γνώμη τους ότι το ένα είναι το σημαντικότερο, το 5, το 7, δεν ξέρω. Και αναλόγως ε, χαράσσονται οι ε, προτεραιότητες και δεν το κάνω εγώ ως αρχή ας πούμε ο Δήμαρχος ε, λέει πόσα χρήματα υπάρχουν το αποφασίζουν από κοινού και εκτελούνται τα προγράμματα και συμμετέχουν και οι πολίτες γιατί είναι σημαντικό για την καθημερινότητά τους και ξέρουν ποιο είναι το πιο οξύ πρόβλημα και η μεγαλύτερη προτεραιότητα. Ακούσαμε και από τους συναδέλφους διάφορα για προεκλογικές εκστρατείες κτλ. Γιατί μετά ο Δήμαρχος δεν ε, έρχεται να λογοδοτήσει υποτύπων εδωλίου, ε, ε, αλλά μπορεί να επικαλεστεί τη συμμετοχή των ίδιων των δημοτών στις αποφάσεις. Κλούζ είναι η πόλη αυτή στη Ρουμανία. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες πόλεις, το Σαν Φρανσίσκο ή το Βερολίνο που συμμετέχουν οι δημότες. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Να ρωτάμε τους πολίτες, τι θέλετε να κάνω ως δήμαρχος, ποια είναι η προτεραιότητα του λαού της πόλης. Δεν κάθομαι σε ένα γυάλινο πύργο να αποφασίζω. Συμμετέχουν και οι πολίτες. Ευχαριστώ. Ε, μια στιγμή, ε, ξέχασα να πω για τις τροπολογίες. Όλοι θέλουμε να είναι καλή η έκθεση και σημαντική και χρήσιμη. Ε, ε πολιτική συνοχή να είναι καλύτερη και να φαίνεται, να προβάλλεται καλύτερα. Περιμένω τις τροπολογίες σας λοιπόν. Άλλο συνάδελφο. Παρακαλώ, κύριο Σχέτμαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια πρόταση, αν μου επιτρέπετε, να πω στο τέλος αυτής της συζήτησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπούντα για την έκθεσή του. Και αυτά που αναφέρεται είναι εξαιρετικά κρίσιμα για την προβολή και την ε, προώθηση της πολιτικής συνοχής, για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα διάφορα έργα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα. Θέλω όμως να τονίσω δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία σε αυτές τις δραστηριότητες προβολής και διαφήμισης. Είναι γεγονό ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν γνωρίζουν πολύ τι είναι η πολιτική συνοχής. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Και στην Πολωνία είναι πολύ ψηλότερο. Αλλά Κατά παράδοξο τρόπο, ακόμα και αν 70% των Πολωνών γνωρίζουν τι είναι η πολιτική συνοχή και τι αποτελέσματα έχει, δεν σημαίνει ότι είναι καλή η κατάσταση και ρόδινη. Και έχουν ε, υποστεί και μία κόποση. Ε, υπάρχει υπερπροβολή στην Πολωνία και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ότι σε κάποια κράτη-μέλη ε, πρέπει να απαντήσουμε στους λαϊκιστές και ε, ο ένας ε, τρόπος είναι βεβαίω να παρουσιάσουμε σωστά αυτά που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο ευρωενθουσιασμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να συνδέεται μόνο ε, με τα κονδύλια που παίρνουμε ε, και τις επιδοτήσεις. Πρέπει να κερδίσουμε και την καρδιά και το μυαλό των πολιτών μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πείραμα, είναι ένα εγχείρημα, είναι ακόμα εν εξελίξη. Και αν μου επιτρέψετε να προβοκάρω λίγο στο τέλος, εγώ θα επιθυμούσα να αλλάξουμε το δόγμα που είχαμε στο παρελθόν για την προβολή ε, της ε, πολιτικής συνοχής. Χρειάζεται να δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία. και να απαγορεύσουμε όλες αυτές τις πινακίδες με τα αστεράκια, με τις σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διάφορα διαφημιστικά γκάτζετ που έχουμε, φλιτζάνια για τον καφέ, στυλό και δεν συμμαζεύεται. Ας δούμε τι συμβαίνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις πολιτικές μας ομάδες. Βγάζουμε συνέχεια τέτοια γκάτζετ σε απίστευτα ε, νούμερα, σε ποσότητες. Αν θέλουμε να αγγίξουμε του πολίτε, χρειάζεται μεγαλύτερη φιλοδοξία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν μέχρι και κατευθυντήριε γραμμέ για τον τρόπο με τον οποίο θα προβάλλει ένα έργο ο δικαιούχο. Και οι κατευθυντήριε γραμμέ, λοιπόν αυτέ λέγουν ότι πρέπει να βάλει συγκεκριμένη πινακίδα με συγκεκριμένες διατάξεις στο έργο. Δηλαδή μέχρι εκεί φτάνουν οι κατευθυντήριες γραμμές και το μέγεθος των ε, χαρακτήρων ε, στη πινακίδα. Σου αφαιρεί όλη τη χαρά της διαφήμισης αν είναι πια τόσο σχολαστική η κατευθυντήρια γραμμή. Ε, Μάλιστα. Όπως γνωρίζετε, η ψηφοφορία προβλέπεται για τον Μάιο και 28 Μαρτίου το μεσημέρι στις 12 είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Όπως ξέρετε, χτες λάβαμε τα πρακτικά της συνεδρίας των συντονιστών, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις θεωρούμε πως εγκρίνονται. Μάλιστα. Θεωρούμε λοιπόν ότι έτσι κλείνει η... Μάλλον υπάρχει κάτι για τα διάφορα, όχι. Οπότε, τέλος της συνεδρίας σας. Ευχαριστώ.